στον κανονισμό. Σας ευχαριστώ. Τα πρακτικά τώρα της ε, συνεδρίας 18 Σεπτεμβρίου είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι, ωραία, εγκρίνονται.